η προθεσμία από αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή από αύριο 21 Ιανουαρίου. Τα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρχή της επομένης περίοδου συνόδου. Εάν δεν έχετε ενστάσεις, τα σχετικά κείμενα θα διαβιβαστούν στους παραλήπτες τους των ψηφισμάτων δηλαδή. Ο κ. Στέρλινγκ, μόλις κάναμε δύο ονομαστικές ψηφοφορίες κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί είχαμε μόνο δύο ονομαστικές ψηφοφορίες. Θα πρέπει να ψηφίζει κανείς άνω του 50% του χρόνου και άνω του 50% των ε, ονομαστικών ε, ψηφοφοριών ώστε να μπορέσει κανείς να λάβει την ημερήσια αποζημίωση. Συμβαίνει αυτό στην παρούσα περίπτωση. Ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να είστε παρόν στο 50% του χρόνου. Συνεχίζει ο Πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, λίγη η σημερινή συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και καλή επιστροφή στα σπίτια σας.